It's just like for, Colleagues. Συνάδελφοι. First of all, my apologies for being a little late. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα κάπως. Μάλλον θα έπρεπε να παραιτηθώ για το λόγο αυτό. Έχετε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι με το σχέδιο ημερήσεις διάταξη. Ωραία. Καταρχάς ε, να καλωσορίσω ε, προσκεκλημένους από την κάτω Σαξονία που βρίσκονται εδώ κατόπιν πρόσκλησης της κυρίας Μάισνερ και επίσης μου είπαν ότι μεταξύ αυτών ε, των τριών κυριών των τριών νεαρών κυριών που μπορεί στο μέλλον να είναι πολιτικοί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα στο μέλλον να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία εάν ε, ακολουθήσετε το όνειρο αυτό. Χαιρόμαστε πάντως που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών. τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών. Ε, θα είμαι σύντομος. Είχαμε μία παρουσίαση από την Γενική Διεύθυνση ε, για τις ε, μεταφορές σχετικά με τον κατάλογο αεροπορικών γραμμών που απαγορεύεται να λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η λεγόμενη μαύρη λίστα. Δεν θέλω να τη λέμε έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται. Οι συντονιστές λοιπόν σημείωσαν τις πληροφορίες που τους δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης ε, σημειώσαμε τα ενημερωτικά σχετικά με την επιτροπολογία υπαριθμών 10, 11 και 12 που εκδόθηκαν τον Μάρτιο και ακούσαμε και την αναφορά της κυρίας Γκρός σχετικά με την αποστολή στη Μαδέρα που νομίζω ότι ήταν πολύ πετυχημένη. Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν πάνω σε αυτήν και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γκρός που ηγήθηκε εκ μέρους μου. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρέπει να αλλάξουμε θέση διότι το, μηχάνημα βρίσκεται από αυτή την πλευρά. Στην ε, αίθουσα αυτή που είναι σαν του Αρθούρου τη Τρογγυλή Τράπεζα θα μπορούσαμε παρακαλούμε να ελέγξουμε Ε, να επιτρέψουμε στους προσκεκλημένους από την κάτω Σαξονία να βάλουν και γάλα στο τσάι τους και τα αποτελέσματα θα τα βλέπετε μόνο μπροστά σας. Δεν έχουμε μεγάλη οθόνη που να δείχνει τα αποτελέσματα σήμερα, εντάξει. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι στη δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Έγκριση της συμφωνίας ε, με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάνω σε μια πρόταση οδηγίας για την ε, χρήση εναλλακτικών καυσίμων, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Έπρεπε βέβαια να αναφέρω ότι είναι έκθεση του κυρίου Φιντάντσα. 28 υπέρ, 2 κατά, 2 εποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Φιντάντσα. Είναι παρόν ο Κάρλο. <laughs> Πολύ δημοφιλής ο Κάρλο. Κατόπιν έχουμε πρόταση μάλλον έγκριση της συμφωνίας με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για ε, ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η συγγήτρια είναι η Γκεζίνε Μάισνερ, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι λήξη της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 4 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ. Gesine, did you want to say a word after this? Gesine, θέλεις ε, να πεις ε, δύο λόγια μετά την ψηφοφορία αυτήν. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Ναι, βέρδεψα τα κουμπιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, διότι ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία μας. Ε, πράγματι δεν πίστευα ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα και το ότι τελικά τα καταφέραμε οφείλεται στην καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, με τον Βέρνερ, τον Κίθ και τον Σπύρο, που με βοήθησαν να κάνουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις. Ε, το Συμβούλιο επέμενε ε, στα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν τώρα γαλάζια ανάπτυξη με ελεγχόμενη ανάπτυξη. Θέλουμε οι θάλασσες να παραμείνουν υγιείς. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Thank you Ευχαριστώ. Κατόπιν θα ψηφίσουμε πάνω στην συμφωνία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την χρήση του συστήματος e-call. Ε, ε, η συγκρίση είναι ο Φιλίπ Τεπάκερ, αρχή της ψηφοφορίας. everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Νομίζω μόλις είδαμε ότι θαύματα γίνονται. 23 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ντεμπάκερ. Πρωτού να προχωρήσουμε, έχουμε την οικογενειακή φωτογραφία για την έκθεση. Θα παρακαλούσα τους βουλευτές ε, να προσέλθουν στο κέντρο της αίθουσας για να τραβήξουμε τη φωτογραφία πρωτού προχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι παρακαλώ κάντε λίγη υπομονή. <laughs> <laughs> Ο πρόεδρος θα φορέσει και τη γραβάτα του, προσέξτε με.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 Η φωτογραφία θα συμπεριληφθεί στην πενταετή έκθεση της Επιτροπής μας. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσετε να πάρετε δικά σας αντίτυπα αν θέλετε. Πάντως θα συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η φωτογραφία. Και έτσι την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσετε να πάρετε και την έκθεση της τελευταίας πενταετίας της, έκθεσης, ε, της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού. Είναι πολύ καλή έκθεση αυτή, έχει και τις φωτογραφίες σας. Ε, η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι σε κάθε έκθεση έχουμε και φωτογραφία του εισηγητή. Πάντως θα είναι έτοιμη η έκθεση αυτή την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι περιορισμοί θορύβου στους Αερολιμένε της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ένα λεπτό να πιούμε και λίγο τσάι. Είναι έκθεση του Γιώργ Λάιχτφριντ. Ο Γιώργ δεν είναι παρόν σήμερα, γι' αυτό θα σας ε, διαβάσω το σημείωμα που μου ετοίμασε. Έχει ως εξής. Ο εισηγητής επικροτεί την θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση που αντικατοπτρίζει την ε, συμφωνία που επιτεύχθηκε στους τριμερείς διαλόγους και που εγκρίθηκε επίσημα από την Επιτροπή ε, Μεταφορών στις 11 Φεβρουαρίου του 2014. Ο εισηγητής είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, διότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να διατηρήσει πολλές σημαντικές ρήτρες, όπως είναι οι πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, ο μετριασμός των ε, ε, των λαβερών συνεπιών για την υγεία των ε, πολιτών θα αναφέρεται ως ε, σημαντικό στοιχείο του κανονισμού. Επίσης αναφέρεται η αναθεώρηση του, της οδηγίας για τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και συμπεριλαμβάνεται και παραπομπή στην οδηγία του 2002. Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να φροντίζουν οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους περιορισμούς λειτουργίας θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν, θα πρέπει να είναι προσβάσιμες δηλαδή για τους, ε, κατοίκους που, για τους ανθρώπους που κατοικούν κοντά στα αεροδρόμια και τις αρμόδιες αρχές. Προτού να θεσπιστεί μια, ένας λειτουργικός ε, περιορισμός, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τα άλλα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή μπορεί μέσα σε τρεις μήνες να αναθεωρήσει τη διαδικασία, αν θεωρήσει ότι δεν συνάδει με τους κανόνες. Μπορεί να ενημερώσει την αρμόδια αρχή που θα πρέπει να εξετάσει την κοινοποίηση αυτή τη Κομισιόν και θα πρέπει να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι προθέσει τη ε, προτού εισάγει του λειτουργικού περιορισμού. Οι ε, αρχέ όμω δεν δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, εισαγωγή λειτουργικών περιορισμών που σχετίζονται με το θόρυβο, όπω η απαγόρευση πτήσεων τη νύχτα. Αυτό αντικατοπτρίζει τον στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της επικουρικότητας. Δεδομένου του επιτυχούς αποτελέσματος ε, των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, ο εισηγητής ε, συστήνει στην Επιτροπή να εγκρίνει το κείμενο ως έχει. Επίσης ε, θέλει να τονίσει ότι αν θέλουμε να μείνουμε στην συμφωνία αυτή, θα πρέπει να καταψεφίσουμε πιθανές τροπολογίες. Αυτές λοιπόν είναι οι παρατηρήσεις του κυρίου Λάιχτφριντ. Ε, θέλει κανείς το λόγο, η κυρία Φώστερ. Τζάκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργ που δεν είναι παρόν εδώ σήμερα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στο θέμα αυτό και νομίζω ότι οι συζητήσεις με το Συμβούλιο και με όλους τους ενδιαφερομένους ήταν πολύ επικοδομητικές. Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει στο σωστό συμπέρασμα. Ήταν ε, σημαντικό ε, να συμμορφωθούμε με την ισορροπημένη προσέγγιση φυσικά. ο κάτι που ήδη κάνουμε στην Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σημαντικό θέμα για μας όμως για το κόμμα ECR ε, αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ήταν το θέμα της επικουρικότητας όσον αφορά την υγεία. Τα αεροδρόμια μας, η πολιτική μας, ε, οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις. Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχει λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό, έχουν επιτευχθεί καλές συμφωνίες και συνεχίζουμε να έχουμε παραγωγική και η βιομηχανία αρωματοφορών ε, συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία μας και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Θα συμφωνούσα επίσης ότι δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό τροπολογίες. Ε, γενικά τα κράτη-μέλη μπορούν να εργαστούν με βάση αυτά που έχουν και αν υπάρξουν προβλήματα μπορούν να επανέλθουν. Νομίζω όμως ότι γενικά στο τέλος πετύχαμε καλή συμφωνία. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Εύα Μια σύντομη παρατήρηση. Ο συνάδελφος Λάιχσφριτ πράγματι διαπραγματεύτηκε πολύ καλά. Το αποτέλεσμα σέβεται τις διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τον θόρυβο στα διάφορα αεροδρόμια. Έτσι σέβεται και την αρχή της επικουρικότητα, ε, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για αυτό σκοπό, προκύπτει από τη φύση του θέματος. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις τοπικέ συνθήκες. Την κατεύθυνση των ανέμων, ε, τις βουνοπλαγιές που αντανακλούν τον ήχο κλπ. Γι' αυτό δικαιολογείται εδώ η επικουρικότητα και η σολομενική λύση στην οποία καταλήξαμε όσον αφορά τα δικαιώματα εντός αγωγικών της Κομισιόν ε, πιστεύω ότι είναι καλή. Ένα πρόβλημα παραμένει για μένα, η λεγόμενη ισορροπημένη προσέγγιση. Ξέρω ότι είναι μια διεθνή συμφωνία, αλλά και σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να παρουσιάσουμε επικρίσεις. Ε, κατά τη γνώμη μου ε, είναι πολύ προβληματική βασική αρχή η ισορροπημένη προσέγγιση. Διότι λέει ότι προστασία της υγείας ε, μπορεί να γίνεται όταν είναι, όταν είναι αρκετά φθηνή. Δηλαδή η προστασία της υγείας ε, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο οικονομικό και αν ε, δεν μπορεί να γίνει τότε δεν ε, εφαρμόζεται. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτή τη ισορροπημένη προσέγγιση και ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο θέμα αυτό, διότι τολμώ να προφητεύσω ότι δυστυχώ στο μέλλον θα έχουμε τεράστια προβλήματα σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σε σχέση με την επιβάρηση από το θόρυβο και ε, από τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Okay, Commission. Η Επιτροπή. Εντάχει, ευχαριστώ Πρόεδρε. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Ξέρω ότι είναι δύσκολο σε αυτή την, ε, ε, την αίθουσα. Πρέπει να σας σκανάρω στην ουσία. Η κυρία Μάιστερ. Ε, νομίζω ότι είχε πρώτο το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, ναι, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα του περιορισμού του θορύβου στα αεροδρόμια. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, την υγεία, αλλά θα ήθελα να διαφωνήσω με την Εύα Λίχτενπέργκερ, επειδή με το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα που έχουμε, πιστεύω ότι σεβόμαστε την αρχή αυτή. Είναι σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο και γι' αυτό συμπεριλαμβάνεται. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος όταν έχει κανείς σε μια ισορροπημένη προσέγγιση να ξεχάσει κάποια πτυχή. Αλλά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν επιτρέπει μια τέτοια ερμηνεία. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις πτυχές και την προστασία της υγείας και γιατρικές πτυχές και αυτό είναι καλό. Ακούγεται σαν να έχουμε θεσπίσει ένα νομοθέτημα το οποίο να βλάπτει την υγεία των ανθρώπων. Δεν ήταν αυτό ο σκοπό του Κοινοβουλίου, ούτε πιστεύω ότι είναι τέτοιο το αποτέλεσμα. Ο Ναι. Ο σκιώδης εισηγητής μας ε, δεν είναι σήμερα παρόν. Ε, έχει ε, ανακοινώσει όμως ότι είναι, αποτελεσ... ότι είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Σημαντικό το θέμα για μας ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν διατεθειμένη να βρει έναν συμβιβασμό. Έχουμε καταλάβει, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για το θέμα των αερομεταφορών. Ελπίζω ότι και τα άλλα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο να συνάδουν και αυτά με την ισορροπημένη προσέγγιση. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η συνάδελφος Γκεζίνε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου περιοχή. Στο Λίτιχ έχουμε ε, ε, επενδύσει περίπου ε, ε, ένα εκατομμύριο ευρώ για να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων ε, γύρω από το αεροδρόμιο. Η οικονομία, η οικολογία και η υγεία των ανθρώπων μπορούν να συνδυαστούν και αυτό αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα. Και το θέμα που έχουμε μπροστά μας δεν αποκλείει κάτι τέτοιο, το αντίθετο και γι' αυτό επικροτώ την έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι δυνατόν να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και θα είναι δυνατόν να προστατεύεται στο μέλλον και αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Δεν θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν μας απασχολεί το θέμα και ότι η οικονομία έχει προτεραιότητα σε σχέση με την υγεία των ανθρώπων. Αυτό δεν ισχύει για μας, ούτε στο μέλλον θα ισχύει. Ξέρουμε ότι ο θόρυβος γύρω από τα αεροδρόμια είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και ότι στο παρελθόν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό. Και στο μέλλον λοιπόν θα είναι δυνατόν να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων. Ήθελα να το τονίσω και να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα από την περιοχή μου, όπου έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες στο θέμα αυτό. Εντάξει. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, ο κύριος ε, Λάιχτφριντ ε, έδωσε μεγάλη ε, μάχη και τα κατάφερε και έπρεπε να υποχωρήσουμε σε σχέση με το δικαίωμα ελέγχου των κατεξιοδότηση πράξεων τα μικρά αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Θεωρούμε όμως ε, ότι οι νέοι κανόνες θα εναρμονίσουν τα διάφορα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση τις ε, χρηστές πρακτικές, τις βέλτιστες μάλλον πρακτικές, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συλλογή στοιχείων ε, για τη σωστή λήψη αποφάσεων με βάση επιστημονικά στοιχεία και συγκρίσιμα συνάμα καθώς και την διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο κανονισμός αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή οδηγία και βοηθά τους ανθρώπους να λάβουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με περιορισμούς μέσα στα πλαίσια μιας λύσης κόστους-οφέλους για να περιορίσουμε ε, τα, αρνητικά φαινόμενα, τις αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή πρόκειται για μια εναρμονισμένη ε, ε, διαδικασία, αλλά οι αποφάσεις παραμένουν σε τοπικό επίπεδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να τύχει υποστήριξη από την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο. Προθεσμία 3 Απριλίου, 5 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή στις 10 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα είναι η παρουσίαση εγγράφου εργασίας σχετικά με τα βιοκαύσιμα, με τις συνέπειες της χρήσης τους και ε, η κυρία Μορέλη έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Okay. Thank you. Good morning. Ε, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα πρωταρχικά αποτελέσματα αυτής της ε, μελέτης σε σχέση με την επίπτωση των βιοκαυσίμων στα διάφορα μεταφορικά μέσα που διναργήσαμε το 2013. Ε, πρόκειται για μια συνεκτική μελέτη σε σχέση με τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς και σχετίζεται με όλες τις πτυχές ε, από την ασφάλεια προμήθειας, ε, ε, κλιματικές επιπτώσεις, αλλαγή της χρήσης της γης και πώς τα διάφορα βιοκαύσιμα δρούν μέσα στα πλαίσια στη, τη, συμβατότητας με τις μηχανές και ούτω καθεξής και πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές επιπτώσεις με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Θα είναι σύντομη αυτή η παρουσίαση, γι' αυτό θα σταθώ σε ορισμένες πτυχές, τις πιο σημαντικές που είναι πολύ ε, σαφείς και απλές ως προς τα μηνύματα ως προς την ασφάλεια προμηθείας, προμηθειών είναι ένας από τους πυλώνες των βιοκαυσίμων που συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση των πηγών ε, καυσίμων για τις μεταφορές με χρήση πετρελαίου αλλά και ε, δίζελ. 5,1% αντικαταστάθηκαν το 2011 με βιοκαύσιμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το βιοδίζελ έχει εισαχθεί κατά κύριο λόγο, γιατί δεν έχουμε τόσο υψηλή παραγωγή. Γι' αυτό στα βιοκαύσιμα ε, οπωσδήποτε εξάγουμε ένα μέρος ε, εθανόλης, αλλά δεν ε, μπορούμε να παραγάγουμε το 2020 θα έχουμε εξοικονόμηση 10 ε, δισεκατομμυρίων σε πετρέλαιο και βιοκαύσιμα. Ως προς τις επιπτώσεις της χρήσης, αυτό είναι ένας άλλος βασικός πυλώνας και τα βιοκαύσιμα μπορούν να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, και στις αγροτικές περιοχές, στη γεωργία και στη βιομηχανία καθώς και στα δηληστήρια στην Ευρώπη για τη δημιουργία βιοκαυσίμων. Όμως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι υπάρχει αύξηση φορολόγησης μέσα στα πλαίσια των ε, επιδοτήσεων ή τις υψηλότερες τιμές ε, βιοκαυσίμων. Σε αυτή την περίπτωση οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι η επίπτωση είναι ουδέτερη, αλλά αυτό είναι φυσικό για όλες τις πολιτικές, διότι όταν υπάρχουν ε, παράπλευρες συνέπειες όπως ε, η υψηλότερη φορολόγηση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό επηρεάζει και τα βιοκαύσιμα. Πόσο μας στοιχίζει αυτή η πολιτική υπέρ των ε, βιοκαυσίμων και πόσο μας στοιχίζει η επιδότηση. Όπως ξέρετε, επιδοτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα βιοκαύσιμα και το κόστος είναι το 2011 7 έως 8,4 δις ευρώ, δηλαδή 14 με 17 ευρώ ανά άτομο, εξαρτάται από τις μελέτες. Από πού προέρχεται αυτό το επιπρόσθετο κόστος. Προέρχεται από το υψηλότερο κόστος παραγωγής, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα ορυκτά καύσιμα έχουν χαμηλότερο κόστος. Μιλάμε λοιπόν για ένα 67%. Αυτό είναι το κόστος παραγωγής. Ε, ως προς τα βιοκαύσιμα σε σχέση με τα ορικά, ορυκτά καύσιμα. Και αυτό οφείλεται στο κόστος ε, πρόσμιξης ή ε, διοικητικό κόστος. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά το κόστος παραγωγής. Μπορούμε όμως να, μιλώ, να μειώσουμε τις τιμές βιοκαυσίμων έτσι ώστε να εξισωθούν με τα ορυκτά καύσιμα. Ως προς τις επιπτώσεις στη γεωργία, βεβαίως ξέρουμε ότι θα πρέπει να γίνει λόγος για το βιοντίζελ και φυσικά ε, αυτό οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης φυτικών ελαίων και το ίμιση της αυξανόμενης ε, ε, ζήτησης αφορά ε, ιδιαίτερα το φινικέλαιο, τις εισαγωγές και ιδιαίτερα του φινικελαίου, κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις ε, στις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, διότι το φινικέλαιο ε, παράγεται στην ε, Μαλαισία και την Ινδονησία σε γη από κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις ε, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα εξαιτίας της διαδικασίας άρδευσης που χρησιμοποιείται. Επίσης χρησιμοποιούμε ένα πολύ μικρό μέρος φινικελαίου για τα βιοκαύσιμα και το μεγαλύτερο ε, αφορά την χρήση άλλων ελαίων όπως της ε, ελαιοκράμβης. Ως προς την εθανόλη τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυσκολότερο να δούμε τις επιπτώσεις της αυξανόμενης ζήτησης στην παγκόσμια αγορά, γιατί η αγορά σιτηρών είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά εθανόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ μεγαλύτερη από την αγορά ε, ελαίων, φυτικών ελαίων. Άρα, για να δούμε την επίπτωση ε, εθανόλης ε, στα δημητριακά, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε απτά αποτελέσματα, διότι τα μοντέλα, τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε είναι διαφορετικά και η αγορά εθανόλης στην Ευρώπη είναι σχετικά μικρή. Άρα η αγορά είναι μικρή διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούμε λιγότερη εθανόλη από βιοκαύσιμα. Ε, και αυτό είναι κάτι που αποτελεί ένα θέμα ίσονος σημασίας. Εδώ στο, στη γραφική παράσταση βλέπετε τις ε, τιμές που έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τον ε, πληθωρισμό των ε, φινικελαίων του Φινικελαίου ιδιαίτερα, ε, μέχρι το 2011 στη ε, μαύρη γραμμή είναι το αργό πετρέλαιο. Βλέπετε από αυτή τη γραφική παράσταση από το 1980 στο 2005 που βλέπετε με την μπλε, ε, στο μπλε γράφημα, οι τιμές των Δημητριακών δεν σχετίζονταν καθόλου με τις τιμές αργού πετρελαίου και οι τιμές έπεφταν διαχρονικά από το 1980 μέχρι το 2005. Το 2005 όπου ε, εμφανίστηκαν και τα βιοκαύσιμα βλέπετε ότι αντιστρέφεται αυτή η τάση, δηλαδή υπάρχει μια ανωδική τάση των ε, τιμών, ιδιαίτερα για τις ζωοτροφές που σχετίζονται βεβαίως και με το αργό πετρέλαιο. Υπάρχει λοιπόν ένας συσχετισμός της εισόδου των βιοκαυσίων με το αργό πετρέλαιο και τις ζωοτροφές. Εδώ βλέπουμε ιδιαίτερα με τον αραβόσιτο στις ζωοτροφές ότι υπάρχει συσχετισμός με την τιμή αργού πετρελαίου και δηλαδή αντιστρέφεται η φθήνουσα αυτή πορεία που γνωρίσαμε μέχρι το 2005. σε σχέση με τις εξοικονομήσεις της εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Αυτό το θέμα συζητήθηκε τα δύο-τρία τελευταία χρόνια ε, εξαιτίας της ε, αλλαγής χρήσης της γης, έμεσης αλλαγής χρήσης της γης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να οδηγούν σε εξοικονομήσεις ιδιαίτερα αν δούμε την τιμή παραγωγής καλλιέργειας και μεταφοράς. Ε, κρίνουμε λοιπόν ότι το 2011 24.000 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα εξοικονομήθηκαν γιατί τα βιοκαύσιμα είναι πολύ υψηλότερα από τη χρήση εθανόλη στην Ευρώπη. Εάν συμπεριλάβουμε σε αυτόν τον υπολογισμό τις εκπομπές με βάση την έμεση αλλαγή χρήσης της γης, το iLook, για τα βιοκαύσιμα βλέπουμε ότι δεν γίνεται εξοικονόμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα σας εξηγήσω αυτές τις εξοικονομήσεις για να σας πω πώς μπορούμε να ε, εξοικονομήσουμε σε εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Ε, ε, βλέπετε ότι το, το γαλάζιο είναι ο, ο κύκλος εκπομπών και αριστερά έχετε την εθανόλη και τις ζωοτροφές ενώ δεξιά έχετε τα βιοκαύσιμα. Εδώ βλέπετε την ποσοστή αναλογία ε, εξοικονόμησης με βάση ε, τα βιοκαύσιμα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν για το ζαχαροκάλεμο και για τα ζαχαρότευτλα βλέπετε ότι γίνονται εξοικονομήσεις ενώ είναι χαμηλότερες για τον ε, αραβόσιτο και τα δημητριακά. Για το άχυρο, όσο αφορά το άχυρο, βλέπουμε ότι γίνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση εκπομπών. Αλλά το σκούρο μπλε ε, είναι το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται και το iLook. Αλλά ιδιαίτερα για τα βιοκαύσιμα έχετε αύξηση εκπομπών, άρα ε, η επίπτωση iLook είναι σχετικά υψηλή σα είπα όμως ότι υπάρχει δυνατότητα για μείωση εκπομπών θερμοκηπίου. Τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να μειώσουμε τον ε, κύκλο ζωής εκπομπών θερμοκηπίου αν χρησιμοποιήσουμε τα παράπλευρα προϊόντα για να, οδηγήσουμε, για να ε, τα χρησιμοποιήσουμε για άλλες χρήσεις, γιατί πάντα υπάρχει ένα υποπροϊόν από τη χρήση βιοκαυσίμων και μπορείτε να το κάψετε και να χρησιμοποιήσετε την, ε, το χρησιμοποιήσετε ως πηγή θέρμανσης. Είτε πρόκειται για ε, δημητριακά ραβόσιτο ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, τα υποπροϊόντα χρησιμοποιούνται και ως ζωοτροφές. Και έτσι χάνουμε και τα δικαιώματα χρήσης υποπροϊόντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ως προς την ε, καλλιέργεια τύρφης, μπορούμε να έχουμε μείωση ε, αυτών των ε, εκπομπών εάν γίνεται καλλιέργεια επί της, επί της γης όπου υπάρχει τύρφη και έτσι θα μειωθεί η έμεση αλληλεγγύη χρήση της γης. Και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση και ως προς το, τα βιοκαύσιμα. Επίσης, στην εγκαταλειμμένη γη μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση και όλα αυτά με τη χρήση βιοκαυσίμων μπορούν να μειώσουν την, ε, τις εκπομπές iLook. Το κόστος τώρα των ε, των εξοικονομήσεων από διοξίδιο του άνθρακα. Το βλέπουμε ιδιαίτερα Ω προ τι μεταφορές όπου το κόστος είναι πολύ υψηλό σε σχέση με άλλες μεθόδους, όμως έχει μεγάλη σημασία και για το τομέα των μεταφορών. Με βάση τα στοιχεία για τις εκπομπές αερίων ε, θερμοκηπίου και το κόστος ε, παραγωγής ε, βιοκαυσίμων, κρίνουμε ότι υπάρχει εξοικονόμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, όπως βλέπετε εδώ, μετά από και επειδή αυξάνονται οι εκπομπές πολλές φορές το κόστος είναι πολύ υψηλό. Να περάσω τώρα στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται με αυτά τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Σίγουρα είναι πολλά υποσχόμενα για τις οικονομίες αερίων του θερμοκηπίου Υπό τον όρο όμω ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις και οι οικονομικές και οι περιβαλλοντικές προκειμένου να γίνει πλήρης ε, απολογισμός του πραγματικού αντικτύπου των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Για παράδειγμα, και τώρα και στο μέλλον θα, χρησιμο... θα ε, απαφεθούμε στην δασοκομεία για τη χρήση γης, αλλά η ουδετερότητα του άνθρακα για τη χρήση δασών για τη βιονέργεια δεν είναι ε, σίγουρο στοιχείο και ιδιαίτερα αν χρησιμοποιήσουμε ε, το, τον κορμό των δέντρων, το βασικό τμήμα της, ε, του δάσους δηλαδή για τα βιοκαύσιμα. Επίσης, ε, τι γίνεται με τη χρήση των υπολείπων ή των αποβλήτων. Με αυτή τη χρήση θα έχουμε ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα. Τώρα, τι γίνεται με το χρήση του αχύρου. Μερικές φορές χρησιμοποιεί θεωρείται ως μηδενικό το παράδειγμα. Δεν είναι μηδενικό, είναι μικρό αλλά όχι μελιτέο. Θα πρέπει όμως και αυτό να ληφθεί υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτροπή αποβλήτων και υπολείπων, που είναι η πιο πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη δεύτερη γενιά των βιοκαυσίμων. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα των ε, συγκεκριμένων τρεχούσων χρήσεων. Αν κάνουμε μία ανάλυση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς θα πρέπει να δούμε το βασικό σενάριο που είναι η χρήση, ε, υπάρχουσα χρήση των υλικών. Θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα της ε, απομάκρυσης, δηλαδή ε, συνήθως το άχυρο μένει στο έδαφος. Τι αποτελέσματα θα έχουμε αν αφαιρέσουμε το άχυρο από το έδαφος. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί το έδαφος ε, και μπορεί η περιεκτικότητα του άνθρακα να μειωθεί και αυτό θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης να δούμε τι γίνεται με το αποτέλεσμα της μετατόπισης γιατί ήδη έχουμε συγκεκριμένη χρήση αυτών των, ε, πρώτων, των ε, ζωοτροφών ή των βοσκοπτόπων. Τι θα γίνει αν χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και με, τέτοιο συνυπολογισμό έχουμε μεγάλες οικονομίες ε, για τα δεύτερα γένια, για τη βιομηθάνη από τη βιο, ε, βιο, ε, χώνευση. εδώ και αν λάβουμε υπόψη κάποια τεχνολογικά στοιχεία, όπως την αφήνοντας τελειπάσματα μετά την παραγωγή της βιομεθάνης, Έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, οικονομίες, αλλά η παραγωγή τέτοιων βιοκαυσίμων εξακολουθεί να είναι αρκετά δαπανηρή. Οπότε η πρόοδος για τα καύσιμα δεύτερης γενιάς είναι πιο αργή από ό,τι από το αναμενόμενο, αλλά έχουμε υψηλό κόστος ακόμη. Έχουμε τεχνολογίες, θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να μειώσουμε το κόστος και να βρούμε τρόπο να εξασφαλίσουμε φτηνές ζωοτροφές και να αναβαθμίσουμε τις διαδικασίες. Με βάση υπολογισμού τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργεια, τα βιοκαύσιμα δεύτερη γενιά σε σχέση με τα βιοκαύσιμα πρώτη γενιά για την περίοδο 2026 μέχρι 2050 και ανάλογα με, τα, με τις τιμές του πετρελαίου ε, θα έχουν πολύ μεγαλύτερη οικονομία. Τώρα, σε σχέση με τα ε, βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς, από φύκια για παράδειγμα, είναι κάπω πρόωρο να κάνουμε υπολογισμού γιατί δεν θα έχουμε εμπορική του χρήση. Είμαστε ακόμη σε φάση έρευνας και τεχνολογική ανάπτυξη για τα βιοκαύσιμα από φύκια. Πάντως όλοι οι οικονομικοί τελεστές ε, ζητούν και απαιτούν σταθερό πλαίσιο, σταθερή πολιτική και σαφή ενάψματα για να συνεχίσουν την, ε, τις έρευνες και την ανάπτυξη των ε, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Και έρχομαι τώρα στα συμπεράσματά μου διαπιστώσαμε ότι τα βιοκαύσιμα είναι μία από τις ελάχιστες επιλογές που έχουμε για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων στον τομέα των μεταφορών, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο. Το βιοκαύσιμο, ε, τα βιοκαύσιμα είναι ακριβή επιλογή και είναι μία από τις ελάχιστες επιλογές που έχουμε, οπότε είναι ακριβή επιλογή για την ε, εξοικονόμηση καυσαερίων σε σχέση με άλλες χρήσεις. Οπότε σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο φθηνό να εξοικονομήσουμε καυσαέρι καίγοντας ε, ε, κάποιες, ε, κάποια, κάποιες για να παράγουμε ενέργεια από το να τα μετατρέψουμε σε βιοκαύσιμα. Τώρα, δεδομένων των περιβαλλοντικών ανησυχιών που δημιουργήθηκαν για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, διαπιστώσαμε την ανάγκη επιτάχυσης της ε, προσπάθειες για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Και αυτή είναι η προσέγγιση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως ε, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα αποτελέσματα της ε, χρήσης και της κατασκευής βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και από απόβλητα κατάλοιπα και το καθεξής. Πάντως θα πρέπει η μετάβαση αυτή να επιταχυνθεί να ληφθούν υπόψη όμως όλες οι επιπτώσεις και ο ανταγωνισμός σχέση με άλλους τομείς και όλες οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν τώρα η οικονομική αποδοτικότητα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Θα πρέπει καταρχήν να έχουμε πρόσβαση σε φθηνές πηγές ε, βιώσιμων ε, βοσκοτόπων και βιοτροφών και φυσικά θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι τεχνολογίες για την παρασκευή τέτοιων βιοκαυσίμων. Ε, χρηματοδοτούνται ήδη πολλά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, το NER 300 είναι ένα από τα πιο μεγαλεπίβολα προγράμματα που χρηματοδοτεί την έρευνα σε προωθημένες μορφές βιοενέργειας. Επίσης, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χρηματοδοτεί την έρευνα για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Πιστεύω με όλες αυτές τις προσπάθειες να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Έχουμε φυσικά και έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης. Εκεί θα καλύψουμε όλες τις πτυχές των βιοκαυσίμων δεύτερη και τρίτη γενιάς. Σας ευχαριστώ και περιμένουμε με αδημονία τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας επί της μελέτης μας, ώστε να, την οριστικοποιήσουμε την έκθεσή μας. Βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού η έκθεση, σε φάση εκπόνηση, γιατί περιμένουμε τα σχόλια της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρός, η κυρία Μάισνερ και η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Όποιος άλλος παρακαλώ επιθυμεί να μιλήσει, να το δηλώσει για να τον περιλάβω στον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή της μελέτης αυτής. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να μειώσουμε <clears throat> τις διάφορες πληροφορίες. Ήθελα να πω όμως κάτι που σχετίζεται με αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε την ε, δυνατότητα να εξετάσουμε την τρίτη γενιά βιοκαυσίμων, τα μικροφύκια, και πιστεύω ότι αξίζει να προσέξουμε το πρόγραμμα αυτό. Πιστεύω ότι θα έχει σημασία για το μέλλον. Διότι ήδη έχουμε περάσει την πρώτη φάση ερευνών, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να παραχθεί πολύ οξυγόνο από τα αφήκια και να έχουμε ένα προϊόν 100% φυσικό, το οποίο να έχει και όλες τις θετικές ιδιότητες του πετρελαίου. Από τη μία τα βιοκαύσιμα αναφέρονται σε ένα πολύ βασικό φαινόμενο της φύσης. Δεν επιβαρύνεται η φύση για την παραγωγή αυτών των καυσίμων ε, και τρίτον ε, μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στην, ε, στο τέλος της παρουσίασής σας στην τρίτη γενιά βιοκαυσίμων. Εσείς πώς βλέπετε προσωπικά τις εξελίξεις αυτές και όσον αφορά τον τομέα των ερευνών, αλλά και στην συνέχεια στους διάφορους τομείς. Υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις όσον αφορά την... Ε, μάλλον υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα στη θάλασσα, η υψηλή θερμοκρασία, ε, ο ήλιος. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν καλές δυνατότητες ε, να προωθηθούν αυτά τα βιοκαύσιμα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, ε, από στενά τις εξελίξεις, ε, να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις αυτές στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη μελέτη αυτή. Την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν έχουμε συνεννοηθεί, αλλά όπως και ο κύριος Γκρός θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στα φύκια, στην τρίτη γενιά βιοκαυσίμων. Θέλουμε να μειώσουμε ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στις μεταφορές. Έχουμε δει πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Ε, τα βιοκαύσιμα λοιπόν ε, δεν είναι εξορισμού βιώσιμα και χρήσιμα για το περιβάλλον και για μας. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην καλλιέργεια τροφίμων και καυσίμων. Θα πρέπει λοιπόν να το θυμόμαστε αυτό. Πριν από δύο χρόνια ε, είδα μία παρουσίαση στην Airbus ε, σχετικά με τα αεροπλάνα του μέλλοντος ε, και μου είχαν πει ότι το καύσιμο είναι τα φύκια. Φαίνεται λοιπόν πολύ φιλικό προς το περιβάλλον αυτό, διότι μπορούν με υδάτινες καλλιέργειες να παραχθούν τα φύκια και μάλιστα σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν δεν κλέβουμε γη από τις άλλες καλλιέργειες. Εσείς πόσο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα βιοκαύσιμα και η δεύτερη με ερώτηση είναι ποιοι θα λάβουν τη μελέτη αυτή, ποιοι θα λάβουν τις πληροφορίες αυτές και θα υπάρξουν συνέπειες για την ευρωπαϊκή πολιτική από τη μελέτη αυτή. Ευχαριστώ κύριε Λίχτενμπέργκερ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και εγώ θεωρώ την έκθεση αυτή πολύ σημαντική στην συζήτηση που μπορούμε να μειώσουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές. Κάποια από τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά. Το γεγονός δηλαδή ότι εμείς εισάγουμε ε, πολύ μεγάλο μέρο των βιοκαυσίμων ε, σίγουρα δεν ήταν ε, ο στόχος. Δηλαδή ότι εμεί ουσιαστικά επιβαρύνουμε τα δάση του Αμαζονίου. Δεν είναι αυτό ο στόχο της χρήση των βιοκαυσίμων. Και υπάρχει και ο ανταγωνισμός με την καλλιέργεια τροφίμων, αλλά και αλλά και η η υπερβολική εκμετάλλευση των δασών ε, του Αμαζονίου επίσης ε, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Εκπρόσωπος ε, Βραζιλιάνων καλλιεργητών, μου είπε ότι καταβάλλεται προσπάθειες σχετικά με το πώς πρέπει να παράγονται τα βιοκάψιμα, γιατί δεν μας λέτε απλά πώς να τα παράγουμε, να το κάνουμε. Σε αυτό το, με, το μέρος του κόσμου όμως ε, πάντα η καλλιέργεια αυτή είναι εις βάρος ε, των ε, δασών του Αμαζονίου. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια στρατηγική ώστε να μην ζούμε εις βάρος κάποιου που χρειαζόμαστε απαραίτητα, δηλαδή των δασών του Αμαζονίου. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής διότι σίγουρα είναι μια εξέλιξη που προκαλεί ανησυχίες. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ήθελα να ξέρω πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Διότι εάν εισάγεται το 50% και από αυτά μεγάλο μέρος να παράγονται από φοινικέλαιο, τότε έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αυτό είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου. Και επίσης θα με ενδιαφέρει το εξή. Πρόκειται για σημαντικά δεδομένα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η τιμή αγοράς, που είναι ψηλή για τα προϊόντα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Ε, ιδιαίτερα σε νησιά παίζει σημαντικό ρόλο η εισαγωγή παραδοσιακών καυσίμων. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα της τιμής της αγοράς. Και άλλωστε δεν μπορεί ε, να εκτιμηθεί η απώλεια των δασών του Αμαζονίου. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τα καύσιμα δεύτερης γενιάς που είναι πιο αποδοτικά δεν... Τι ποσοστό έχουν στην αγορά και δεν πιστεύετε ότι οι εκτιμήσεις σας για το μέλλον είναι υπερβολικά ε, αισιόδοξε. Υπάρχει υπολογισμός του εξωτερικού κόστους της παραγωγής αυτής. Και επίσης θα με ενδιέφερε γεωγραφικά τι διαφοροποίηση υπάρχει. Πόσο μεγάλο ποσοστό παράγεται στην Ευρώπη, σε περιοχές όπου δεν γίνεται πια καλλιέργεια τροφίμων, τι ποσοστό παράγεται σε ποια άλλα μέρη του κόσμου. Είναι ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες αυτές για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και τα συστήματα επιδότησης στο μέλλον. Ευχαριστώ. κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν σημαντικές ανησυχίες μας και κυρίως ε, η επιφυλάξη μα ω προ τον αντίκτυπο που θα έχει η παραγωγή βιοκαυσίμων στι διάφορε καλλιέργειε. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τα σχόλια των συναδέλφων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα για την έκθεση και αν θα περιλάβετε σε αυτό την ανάλυση του αντικτύπου ε, στις διάφορες πολιτικές των κρατών μελών. Γιατί στα συμπεράσματά σας αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι οι οικονομικοί τελεστές ζητούν σταθερές πολιτικές και σταθερά πλαίσια για να μπορέσουν να αναπτύξουν ε, τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς και όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για όλους τους τομείς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα. Τι αντίκτυπο θα έχει στα κράτη-μέλη η νομοθεσία που θα εφαρμόσουν το καθένα με τον τρόπο του. Είπατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις έρευνες και φυσικά για την πρώτη απαιτείται έρευνα. Μιλήσατε για τα προγράμματα το ορίζοντα 2020, το NER 300 Με βάση τα στοιχεία και τις μελέτες που έχετε κάνει, ε, ποιος κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να πραγματοποιήσει την έρευνα. Να έχουμε πανευρωπαϊκή έρευνα, έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή κάθε χώρα να κάνει την έρευνα μόνη της. Πιστεύω ότι για να έχουμε εναρμονισμένες πολιτικές ε, ε, και για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσετε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο στην απασχόληση, στη γεωργία, στην εκπομπή αερίου του θερμοκηπίου. Πώς κατά τη γνώμη σας θα πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, με ποιο τρόπο, γιατί μία από τις τραγωδίες που βιώνουμε είναι ότι όσες μελέτες και αν έχουμε, όσες εκθέσεις και αν κάνουμε, αν κάθε χώρα εφαρμόζει με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες πολιτικές, εκτός ότι δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε περαιτέρω ανισότητες και ασυμμετρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι δεν θα γίνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα σημείο αναφορά και ένα παράδειγμα προς μίμηση. Οπότε δεν θα σημειώσουμε πρόοδο ούτε στα βιοκαύσιμα τρίτη γενιά, ούτε στη σωστή διάγνωση τη κατάσταση. Εν κατακλείδη λοιπόν, πώ εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη την οδηγία αυτή και τι αντίκτυπο έχει η εφαρμογή της οδηγίας ε, ε, με τη διαφορετική συμπερίληψη της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάνιον. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και είναι αναφυσβήτω ότι η παραγωγή μιας καλλιέργειας και η παραγωγή οποιοδήποτε ε, η παραγωγή βιοκαυσίμου είναι η γέννη δαπανηρή. Είμαι και εγώ παραγωγός βιοκαυσίμου και γνωρίζω ότι ε, με λιγότερο από 70-80 ευρώ τον τόνο δεν μπορεί κανείς να παράγει βιοκαύσιμο από οποιαδήποτε καλλιέργεια. Πάντως τα υγρά καύσιμα είναι ένας δυσεπίλητος τομέας σε ό,τι αφορά την, το στόχο της βιωσιμότητας, της αηφορίας. Οπότε σίγουρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, υγρά καύσιμα για την ε, θέρμανση, αλλά μόνο θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε εκεί που είναι απολύτως απαραίτητα, γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, βιώσιμη λύση. Επίσης, το κόστος της βιεθανόλης από δημητριακά, κυρίως από ΣΥΤΟ, τεράστιο το κόστος. Και παρακολούθησα κάποιες έρευνες που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα πορίσματα τους λένε ότι το κόστος ε, οικονόμησης ε, των καυσαερίων από χρήση ε, εθανόλης από σίτο και από ζαχαροκάλαμα ή και ζαχαρότευλο και ο υπολογισμό του εξαρτάται από την μέθοδο που χρησιμοποιείται γιατί ε, η βιεθανόλη είναι ε, τρόφιμο υψηλής πρωτεΐνης οπότε έχουμε μεγάλο συμπίκνωμα πρωτεΐνης που θα μας ε, επιτρέψει να εισαγάγουμε πολύ λιγότερη σόγια από τη Βραζιλία και από τα τροπικά της δάση. Οπότε αν και τέτοιοι παράγοντες υπόψη οικονομία των καυσερίων είναι πολύ ψηλότερη και το αποτέλεσμα που μας δίνει η έρευνα είναι πολύ καλύτερο. Αρκεί να ληφθούν υπόψη και αυτοί οι παράγοντες που προανέφερα. Επίσης, για τις αζωτούχες ενώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εσοδεία εδώ. Την αναφέρατε κάπως παρεμπιπτόντω. Αν έχουμε υψηλή εσοδεία όμως, θα έχουμε και χαμηλότερες, ε, χαμηλότερους εκπομπών. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως είναι ότι ακόμη και στη χειρότερα σενάρια πολλές φορές ε, εφαρμόζουμε στρατηγικές μετριασμού ιδιαίτερα για τις αζωτούχες ενώσεις και έτσι μπορούμε με τη διαχείριση, με την κατάλληλη διαχείριση, μια και γνωρίζουμε ε, τι προκαλεί τέτοια περιστατικά αζωτούχων ενώσεων, να χρησιμοποιήσουμε στρατηγικές λοιπόν μετριασμού για να μειώσουμε το τμήμα των εκπομπών που προέρχονται από, από αζωτούχες ενώσεις. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αηφορία. Έχουμε πολλούς τρόπους λοιπόν για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια το κόστος της παραγωγής βιομάζας είναι αυτό που θα πρέπει να μειώσουμε πρώτα απ' όλα. πολύ τεχνικά τα θέματα αυτά. Αυτό τα προσπάθησα να αγοβάλω τα ακουστικά μου για να καταλάβω κάτι από τη διερμηνία τουλάχιστον. Ο κύριος Σαβάνα, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνικός και ελπίζω να είμαι και ε, εμπεριστατωμένος. Ελπίζω ε, να μην ε, κρίνουμε όλα τα βιοκαύσιμα εξίσου μη βιώσιμα γιατί αυτά που ακούω εγώ μου φαίνονται μάλλον αισιόδοξα σε σχέση με κάποιες απεσιόδοξες ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το προηγμένα βιοκαύσιμα, ε, οι πρωταγωνιστές της αγοράς ε, μας λένε ότι προβλέπουν να καταρρεύσει η αγορά, η παραγωγή φινικελαίου τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2025. Και ταυτόχρονα αυτό που έχουν ε, αυτοί οι πρωταγωνιστές παγκοσμίω και οι μεγαλύτερες εταιρείες ε, στις ε, προηγμένες τεχνολογίες σε σχέση με τα καύσιμα τρίτης γενιάς, τα αποτελέσματα που έχουν είναι πολύ, πολλά υποσχόμενα και αισιόδοξα. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην συνολική μας προσπάθεια για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως διοξιδίου του άνθρακα, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο βιώσιμη εικόνα παγκοσμίω χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, τις τεχνολογίες εχμής που πραγματικά εξελίσσονται ραγδαία. Και ε, ανά πάση στιγμή, σε 5, 10, το πολύ 15 χρόνια, θα έχουν γενικευτεί και πραγματικά θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Οπότε αυτά που χρειάζονται οι ερευνητές ε, είναι ακριβώς ε, σταθερή νομοθεσία, προβλέψιμη νομοθεσία και πλαίσιο για να έχουν τα ενάυσματα και να μας εξασφαλίσουν σε λίγο χρόνο τις τεχνολογίες εκχμής και τα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, για τη χρήση των δασών. Σίγουρα δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης με τα δάση της Φιλανδίας, της Σουηδίας ή κανένα δύο άλλων χωρών. Αλλά, για παράδειγμα, στην πατρίδα μου έχουμε ε, μειώσει κατά 70% την ετήσια ανάπτυξη. Δηλαδή το 30% της ανάπτυξης ε, πηγαίνει χαμένη. Οπότε, αν αυτό που ακούγεται στους διαδρόμους, δηλαδή το θέμα της βιωσιμότητας για, τη βιομάζα, που θα πρέπει να τύχει διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με την χρήση των δασών, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε φιλικά προς το περιβάλλον, ε, να, το κάνουμε και να το εξορθολογήσουμε, γιατί και εκεί έχουμε πολλές βελτιώσεις να κάνουμε. Γιατί και για το θέμα της δασοκομείας με μερικές φορές παραβλέπουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Κυρία Μαρέλη, θα θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, ε, πληθώρα ερωτήσεων, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον σας για τη μελέτη που πραγματοποιήσαμε να ξεκινήσω με το θέμα των φυκιών. Σίγουρα υπάρχουν πολλές προσδοκίες ε, για την παραγωγή βιοκαυσίμων από φύκια. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν δεν χρησιμοποιείται ε, ε, γη. Επίσης η απόδοση είναι μεγάλη από την παραγωγή φυκιών. Έχουμε ακούσει κάποιες προβλέψεις, δεν υπάρχει ακόμη εμπορία στην αγορά, αλλά μερικοί παραγωγοί μας είπαν ότι μπορούμε να έχουμε και 45.000 λίτρα ανά εκτάριο βιοκαυσίμων, δηλαδή που, που η, ελαίου που παράγεται από φύκια. Επίσης δεν υπάρχει ανταγωνισμός ό,τι αφορά τη χρήση γης. Και από τα φύκια έχουμε και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, οπότε μπορούμε πολλά είδους καύσιμα να παράγουμε από τα φύκια και όχι μόνο βιοκαύσιμα αλλά και ζωοτροφές. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα τα φύκια θα είναι το μέλλον όχι μόνο για τα βιοκαύσιμα αλλά και για πολλούς άλλους τομείς και αγορές. Επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα σε διάφορες φάσεις εξέλιξης για το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε σίγουρα να δηλώσουμε ότι βρίσκονται σε φάση ε, εμπορία, αλλά σίγουρα πολλά ε, προγράμματα βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο. Έχουμε όμως κάποια προβλήματα που θα πρέπει να επιληθούν. Στις τεχνολογίες, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε παραγωγή ε, φυκιών σε ανοιχτές λεκάνες, ανοιχτές δεξαμενές που είναι πιο φθηνό βέβαια, είναι ανοιχτές οι δεξαμενές, οι ανοιχτές οι λεκάνες, αλλά είναι πολύ πιο τροτά τα φύκια από σε εξωτερικούς παράγοντες όταν έχουμε ανοιχτή δεξαμενή. Αλλά είναι φθηνότερη αυτή η λύση από το να έχουμε κλειστή δεξαμενή. Εκεί έχουμε υψηλότερε οδιέ, βρίσκονται στο απειρόβλητο τα φύκια, δεν είναι τόσο ευάλωτα σε εξωτερικά βακτηρίδια ή εξωτερικού άλλου παράγοντε αλλά το κόστος είναι υψηλότερο. Η εσοδία όμως είναι καλύτερη. Η... Τέτοιου είδου όμω φωτοαντιδραστήρε που χρειάζονται για τι κλειστέ δεξαμενέ είναι πολύ δαπανηροί. Οπότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να έχουμε με χαμηλό κόστο δυνατότητα να καλλιεργήσουμε φύκια που δεν θα είναι όμω τροτά και ευάλωτα σε εξωτερικού παράγοντε. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή, αυτή τη στιγμή. Άλλο πλεονέκτημα των φυκιών που αναφέρθηκε από κάποιον προλαλήσαντα είναι ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή ε, για τη χρήση στην αεροπορία και σε άλλους τομείς μεταφορών γιατί για την αεροπορία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε βιοκαύσιμο εξαρτάται ε, από τα χαρακτηριστικά του. Τα φύκια είναι από τα ελάχιστα βιοκαύσιμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην αεροπορία. Οπότε και αυτό είναι πολύ θετικό μεγάλο πλονέκτημα και αυτό των φυκιών. Πάντως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε πότε θα τεθούν σε εμπορία ε, και θα είναι διαθέσιμα σε εμπορική κλίμακα τα φύκια. Γιατί βρισκόμαστε ακόμη στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Και ακόμη και για αυτά τα βιοκαύσιμα οι προβλέψεις μάλλον είναι αισιόδοξε για να μην αναφερθώ στα βιοκαύσιμα τρίτη γενιά, που είναι τα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή το μερίδιο των βιοκαυσίμων δεύτερη γενιά είναι σχετικά χαμηλό. χαμηλό. Είναι κάτω από 1%. Μηδέν και κάτι. Η πρόταση πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο την αύξηση αυτού του μεριδίου βιοκαυσίμων δεύτερη γενιά, προτείνοντα έναν στόχο 2,5% βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών για το 2020. Οπότε δύσκολα θα αυξηθεί αυτό το μερίδιο βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, εκτός και αν δοθούν πραγματικά ισχυρά κίνητρα γιατί το κόστος παραγωγής εξακολουθεί να είναι υψηλό για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Οι τεχνολογίες προχωρούν, οι θερμοχημικές, ε, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που είναι πολλά υποσχόμενες. Ε, τα βιοδηληστήρια επίσης ε, πολύ, πολλά υποσχόμενος κλάδος γιατί δεν ε, παράγουμε μόνο βιοκαύσιμα αλλά και άλλα χημικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς. Πάντως η πρώτη ύλη είναι πολύ ακριβή γιατί για να παράγουμε εθανόλιο από άχυρο. Το άχυρο είναι πάνθινο βέβαια είναι κατάλοιπο ουσιαστικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το άχυρο, να μεταφερθεί στο βιοδηληστήριο που συνήθως βρίσκεται πολύ μακριά από το χωράφι που συνελέγει το άχυρο. Οπότε το κόστος από το άχυρο είναι 68 ευρώ τον τόνο. Πανύψηλο κόστος, σε σχέση με την αρχική τιμή του αχύρου που είναι η πρώτη ύλη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στη Βραζιλία, όπου όλα τα δηληστήρια ε, κατασκευάζονται πολύ κοντά, δίπλα στα χωράφια, δεν έχουν κόστος μεταφοράς για τη μεταφορά του ζαχαροκάλαμου, για παράδειγμα, για την παραγωγή βιομάζας ή βιοκαυσίμου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί με πολύ ε, χαμηλό κόστος χρησιμοποιείται ε, και το, η πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας για, για το ίδιο το δηληστήριο. Γι' αυτό και η, η παραγωγή βιοκαυσίμου από ζαχαροκάλαμο είναι και η πιο φθηνή αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή η, Βραζίλια, η κυβέρνηση της Βραζιλίας δίνει επιδοτήσεις για εθανόλη από ζαχαροκάλαμο. Γιατί ακόμη και με πολύ αποδοτική διαδικασία το η εθανόλη από ζαχαροκάλαμο είναι ακριβότερο και από τη βενζίνη. Ακόμη και στη Βραζιλία που δίνονται επιδοτήσεις για την παραγωγή αυτή. Σε ό,τι αφορά το μερίδιο λοιπόν βιοκαυσίμων δεύτερη γενιά, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Πολύ χαμηλό μερίδιο και αυτέ είναι οι προβλέψει για το μέλλον. Πάντω, δεδομένη παρούσα κατάσταση τη συζήτηση και των εξελίξεων, ίσω ε, οι εξελίξει είναι πιο ραγδαίε, γιατί και οι άλλες πολιτικές αναπτύσσονται προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε με ένα σταθερό πλαίσιο οι οικονομικοί τελεστές θα έχουν πολύ περισσότερα κίνητρα να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Πάντως σας εξήγησα που έχουμε τα προβλήματα και το κόστος των ενζήμων είναι πολύ υψηλό γιατί τα ένζημα είναι απαραίτητα για τη διάσπαση της κυταρίνης, για την παραγωγή της ζάχαρης και άρα της εθανόλης. Οπότε και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, αυτή τη στιγμή εισάγουμε περίπου το 2012 είχαμε εισαγωγή 21-22% των βιοκαυσίμων και 21-22% ποσοστό δηλαδή εισαγωγών εθανόλης. Βέβαια παράγουμε και εσωτερικά ε, βιοκαύσιμα από ελαιοκράμβη, αλλά εισάγουμε μεγάλες ποσότητες φινικελαίου για να αντικαταστήσουμε την ελαιοκράμβη στην παραγωγή βιοκαυσίμου. Οπότε εξαρτόμαστε από τις εμπορικές οραίες και τις εισαγωγές και για τις δύο πρώτες ύλες. Τώρα για, για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς που θα χρησιμοποιούνται από, από που θα παράγονται από απόβλητα ή κατάλοιπα, αυτά θα παράγονται τοπικά, δεν χρειάζεται να τα εισάγουμε δηλαδή. Στην περίπτωση της δασοκομείας όμως ε, ε, εισάγουμε pellets ε, από τη Βόρεια Αμερική. Βέβαια αυτά τα pellets και δεν μιλούμε για, το, για τις μεταφορές, κυρίως για τη θέρμαση κάνουμε τις αγωγές αυτές για θέρμαση και ηλεκτρισμό, αλλά το αναφέρω γιατί είναι πρώτη ύλη τα pellets Επίσης η βιωσιμότητα των pellets γιατί παράγονται από κατάλοιπα της δασοκομείας, αλλά υπάρχουν ενδείξει και κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική, σε μερικές περιοχές νότιο-δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών για παράδειγμα, μία, ένας, ένα, ένα τμήμα της παραγωγής πέλετς γίνεται από ξύλο και όχι από κατάλοιπα ξυλίας ή δασοκομείας. Αλλά είναι σημαντικά τα pellets ε, αυτά, Κυρίω, ε, παραλαμβάνω όχι για τι μεταφορέ, αλλά για τη θέρμανση και τον ηλεκτρισμό. Σε ό,τι αφορά την καταστροφή των τροπικών δασών, το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική είναι σταθερό και στην οδηγία για, τα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ποιότητα των βιοκαυσίμων λέμε ότι σε καμία περίπτωση ε, δεν θέλουμε βιοκαύσιμα που θα προέρχονται από τυρφώνες, από τροπικά δάση. Υπάρχει προστασία δηλαδή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι με τα βιοκαύσιμα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε βιοκαύσιμα που γίνονται από υλοτομία του τροπικού δάσους. Το θέμα, γίνεται, το θέμα προκύπτει με τα μετατόπιση και από την έμεση αλλαγής χρήσης γης. Έχουμε κάποια κριτήρια βιωσιμότητας που είναι σαφέστατα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, αλλά δεν καλύπτονται γιατί έχουμε έμεσα αποτελέσματα, έχουμε μια μετατόπιση. Οι νέε πολιτικές που προτείνονται καλύπτουν και αυτό το σημείο Οπότε προσπαθούμε και εδώ να σημειώσουμε πρόοδο και να μειώσουμε τη χρήση των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς για να μειώσουμε τον αντίκτυπο, τον έμεσο αντίκτυπο στο τροπικό δάσος, πρωτογενές δάσος και στον περιβαλλοντικό κίνδυνο, στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πάντως το 2008 που προτάθηκε η πολιτική ελήφθη αυτό υπόψη, οπότε προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα τροπικά δάση και σίγουρα θέλουμε να προωθήσουμε τα βιοκαύσιμα εις βάρος των τροπικών δασών. Σε σχέση με τη Χέρσαγη, νομίζω ότι έχουν διενεργηθεί μελέτες που είναι υπεραισιόδεξες για την χρήση αυτή της χέρσαγης, διότι υπερεκτιμούν την διαθέσιμη χέρσαγη. Και Με βάση τις στατιστικές του ΦΑΟ που είναι και η πιο αξιόπιστη πηγή δεδομένων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι στατιστικές αυτές ε, της ΦΑΟ θεωρούν ε, τη χέρσαγή και την, ε, τα βοσκοτόπια, τα οποία δεν είναι ε, χέρσαγή, καθαρή χέρσαγή η κτηνοτροφική δηλαδή χρήση επίσης εκεί όπου ε, παράγεται, το στάχι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο ποσοστό της γης των Ηνωμένων ε, Πολιτειών έχει αυτή τη χρήση, δηλαδή ε, καλλιεργείται το στάχι, άρα δεν πρόκειται για χέρσαγη. Σε πολλές ε, περιπτώσεις η εγκαταλειμμένη γη είναι εγκαταλειμμένη διότι η απόδοση είναι πολύ χαμηλότερη από την ε, υπολογιζόμενη ε, στην χώρα αυτή. Άρα η χέρσα γη μας δίνει υπερεκτιμημένες στατιστικές ως προς την σύγκριση του κόστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνώ μαζί σας, αλλά για τα σιτήρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υψηλή ε, παραγωγή και καλά αποτελέσματα. Εμείς δίνουμε ένα μέσο όρο για την Ευρώπη. Γι' αυτό είναι υψηλότερα τα ποσοστά. Ελπίζω να κάλυψα τις, ε, τα περισσότερα ζητήματα. Ε, και στην έρευνα που διενεργείται. Εμείς θέλουμε να επιταχύνουμε, ε, τα στοιχεία, να επιταχύνουμε τη διαδικασία για βιοκαύσιμα τρίτης γενεάς. Και μιλάμε όχι μόνο για πρωτογενή ε, έρευνα, αλλά και μία έρευνα εν του ορίζοντα 2020 όπου αποζητούμε ολοκληρωμένες λύσεις σε επίπεδο κρατών μελών με βάση την πρωτογενή έρευνα, τα βασικά σχέδια επίδειξης γνωρίζοντας ότι δεν χρειαζόμαστε ε, έρευνα αυτή αλλά και επίδειξη, σχέδια επίδειξης ή σχέδια για την αγορά. Άρα ο νέος διαγωνισμός για τον ορίζοντα 2020 θα ασχοληθεί με έρευνα και επίδειξη ε, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ανά κράτος μέλος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ε, σας διακατέχει πάθος, μεγάλο πάθος για αυτό το θέμα και ζέση το ανακτώ. Η γκεζίνε πρέπει να είναι πολύ σύντομη δεν απαντήθηκαν δύο ερωτήσεις μου. Ποιος θα επιβλέψει τη μελέτη το Συμβούλιο και τι ε, επιπτώσεις θα έχει στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως και κάθε μελέτη δημοσιοποιείται όταν ε, ολοκληρωθεί. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, σε μία ε, ενδιάμεση μελέτη. Βεβαίως ε, θα επιβλέψει και το Συμβούλιο. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ε, ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε το Συμβούλιο. Δηλαδή πάντα επιβλέπει και πάντα ασχολείται για την τελική έγκριση. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι εξελισσόμενη και περιμένουμε και σχόλια από τις άλλες γενικές ε, διευθύνσεις. Και σήμερα μάθαμε ότι θεωρείται χέρσα γη εκεί όπου καλλιεργείται το στάχι. Θεωρείται χέρσα γη, ε, εν πάση περιπτώσει έτσι θεωρείται τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και είμαι σίγουρος ότι η νέα Επιτροπή θα ε, λάβει την έκθεση όταν έχει ολοκληρωθεί. Επόμενο θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης ε, Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων. Οι συντονιστές ζήτησαν να αποδοθεί μια έκθεση. Ε, ελπίζαμε ο κύριος Βίνκ να το αναλάβει, αλλά δυστυχώς ο κύριος Βίνκ δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ο κύριος Ρονίνη θα μας πει γιατί στο κέντρο της Ευρώπης αυτό το σχέδιο ε, έχει ε, δεχτεί, έχει, σε αυτό το σχέδιο έχει υπάρξει τέτοια επιβράδυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ο Κάρελ Βίνκ ζητεί καταρχάς συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Παραμένει στη διάθεσή σας όμως για οποιαδήποτε ευκαιρία συζήτησης του θέματος μαζί σας. Είναι προνόμιο για μας να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε λίγα λόγια για την μελέτη πάνω στην εφαρμογή του Σχέδιου Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματο Διαχείριση Κυκλοφορία Σιδηροδρόμων. Κατά τη διάρκεια τη θητεία σα, μα έχετε βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων για να ενισχύσουμε το σύστημα αυτό στην Ευρώπη και να το φέρουμε σε ένα όριμο στάδιο. Μας βοηθήσατε να κατευθύνουμε τα βήματα του ε, Ευρωπαίου Συντονιστή και το ERTMS ε, να είναι ένας ε, βασικός διάδρομος, να το πούμε έτσι, στο νέο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων, Επίσης έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης του ERTMS που ε, προβλέπει κάποιες βασικές διαδρομές να εξοπλιστούν με το σύστημα αυτό. Επίσης, μας έχετε βοηθήσει να εντοπίσουμε τους βασικούς διαδρόμους του ERTMS, καθώς και τους βασικούς διαδρόμους για τα εμπορεύματα, όπου βλέπουμε την μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος. Επίσης, μας βοηθήσατε να ενοποιήσουμε, ε, βρούμε την ευρωπαϊκή υποστήριξη για την εφαρμογή του συστήματος αυτού και τέλος αγωνίζεστε μαζί μας ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων να αποκτήσει περαιτέρω αρμοδιότητες ώστε να μπορέσει να προωθήσει την εφαρμογή του ERTMS σε όλη την Ευρώπη. Το ERTMS είναι σημαντικό για την πραγματοποίηση ε, μιας ενιαίας ευρωπαϊκής περιοχής σιδηροδρόμων. Το βασικό θέμα εδώ είναι η διαλειτουργικότητα. Το ERTMS αποτελεί το βασικό εργαλείο για να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα, αποτελεί όμως και το σημαντικό τεχνικό στοιχείο για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια του δικτύου. Η, η εικόνα που δίνουμε στην έκθεση είναι θετική. Νομίζω ότι το πιο θετικό στοιχείο είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο άνευ επιστροφής όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος αυτού. Ωστόσο και αυτή είναι η κατάσταση που περιγράφουμε και που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε κατακαιρματισμένη εφαρμογή και αναφέρομαι και στην παρατήρηση του Προέδρου. Ιδιαίτερα σε κάποιες κρίσιμες διαδρομές υπάρχει καθυστέρηση εφαρμογής του συστήματος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε το θετικό ότι το ERTMS έχει γίνει όχι μόνο ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά και παγκόσμιο πρότυπο διαλειτουργικότητας και ασφάλειας. Έχουμε 20 κράτη-μέλη σήμερα που χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό. Και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 36 χώρες σε όλον τον κόσμο που εργάζονται πάνω στην εφαρμογή του συστήματος. Αυτό λοιπόν μας θυμίζει τη γενική σημασία για τον τομέα αυτών του συστήματος, διότι στο κάτω-κάτω είναι ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν και στην Ευρώπη και εκτός. Έχουμε λοιπόν την κατακαιρματισμένη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή και Καταρχάς, ε, σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε την ανανεωμένη εντολή που έχετε ε, δώσει στον συντονιστή, τον Κάρελ Βίνκ. Είναι λοιπόν καθήκον του να βελτιστοποιήσει την εφαρμογή, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης. Όποτε εφαρμόζεται το σύστημα, να διασφαλίζεται η ομαλή χρήση του τουλάχιστον στους βασικούς διαδρόμους εμπορευμάτων που έχουν καθοριστεί. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προϋποθέσεις ε, που υπάρχουν ε, στα νέα μέσα χρηματοδότησης. Εσείς ήσασταν βασικοί υποστηρικτές αυτών φροντίσατε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είτε μέσω της χρηματοδότησης για τις έρευνες είτε για περιφερειακά έργα. Φροντίσατε λοιπόν ε, να έχουν σωστές τεχνικές προδιαγραφές τα έργα που χρηματοδοτούνται και να ακολουθούν και την προτεραιότητα όσον αφορά τις διαδρομές ε, τις οποίες θέλουμε να εξοπλίσουμε με το σύστημα αυτό. Τρίτον, ε, θα πρέπει να κάνουμε ε, ένα ριζικό βήμα όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. Όπως περιγράφουμε στην έκθεση, έχουμε ένα μείγμα όσον αφορά την ε, γεωγραφική εφαρμογή και επίσης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. Και δεν υπάρχει λόγος να προωθήσουμε μία λύση εάν τελικά τροποποιηθούν οι προδιαγραφές και έτσι χάσουμε τη βασική αξία που είναι η διαλειτουργικότητα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συντηροδρόμων ώστε να έχουμε φέτος τον Ιούνιο τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ώστε να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Ε, και αυτό σημαίνει και ο βιομηχανικός τομέας και οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας να συγκεντρωθούν ε, στα βασικά στοιχεία ε, του συστήματος, ώστε να εντοπίσουν ποια είναι τα βασικά στοιχεία του συστήματος και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία ωραίο θα ήταν να έχουν, τα οποία να μπορούν να εφαρμόσουν πιο μετά. Ώστε να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης, όσον αφορά την εφαρμογή, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την οικονομική πλευρά της διαλειτουργικότητας. Υπάρχουν ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, ωστόσο θα πρέπει να είναι η οικονομική η εφαρμογή του συστήματος αυτή καθ' αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν καταρχάς να επικεντρωθούμε στα σημεία συμφόρησης, όπως πιστεύω ότι σας εξήγησε και ο Κάρελ Βίνκ όταν σας παρουσίασε την τελευταία του έκθεση. Εάν βρούμε λοιπόν ε, μία λύση ε, σε ένα διασυνοριακό σημείο των διευρωπαϊκών δικτύων θα καλύψουμε το 80% της διασυνοριακής, των διασυνοριακών μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν να καλύψουμε ακριβώς αυτά τα σημεία. Δεύτερον, ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, κάτι που, που αναφέρετε κι εσείς ε, στο πλαίσιο ε, της διευκόλυνσης ε, συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe Facility. Έτσι λοιπόν ε, επιτρέπεται να υπάρχουν πιο οικονομικά δάνεια για την αγορά του ε, εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού. Επίσης, ολοκληρώνουμε την μελέτη αντικτύπου σχετικά με έναν κανόνα εφαρμογής που θα βοηθήσει τους διαχειριστές υποδομής να εφαρμόζουν διαφοροποιημένη τιμολόγηση ώστε να δώσουν κίνητρο για τη χρήση του ERTMS. Και επίσης, Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα διαχειριστών της εφαρμογής, μάλλον στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, για να παράσχουμε υποστήριξη προς τους διαχειριστές για την όσο γίνεται πιο ομαλή εφαρμογή του συστήματος. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Μικρόφωνο δεν ακούμε. Mrs. Lichtenberg is a coordinator, Mrs. Tikal. Okay. Can you try and be as brief as possible? I know. Να είστε σύντομοι, ξέρω ότι θέλει κανείς ε, να υπερβεί το χρόνο του κυρίου Ρονίδη, αλλά θα ήθελα να είσαστε πολύ σύντομοι. Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις πληροφορίες που ακούσαμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι φυσικά το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Είχαμε όμως και πάντα σημαντικές ανησυχίες και νομίζω ότι τις ανησυχίες αυτές τις ημεριζόταν και ο Καρελ Βίνκ που σίγουρα δεν είναι εύκολη η δουλειά του πριν δύο χρόνια έγινε συνάντηση μεταξύ άλλων με την SNCF και την Deutsche Bahn. Και μας είπαν ότι σας παρακαλούμε μην ε, βρίσκεται καινούριο σύστημα κάθε χρόνο, θα πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι έχουμε πετύχει τη σταθερότητα αυτή ή έχουμε ακόμα ένα σύστημα όπου το 2014 θα έχουμε κάποια νέα στοιχεία, το 2015 ε, κάτι νέο και να μην υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στα δύο αυτό. Αυτό για μένα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία. Δεύτερον, ε, το μνημόνιο κατανόησης ε, έχει υπογραφεί. Εγώ θα ήθελα εδώ να δω και κάποιους άλλους εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα παρουσιάζει θετικά μηνύματα, αλλά βλέπω επιφύλαξη από πλευράς ε, των ε, κρατών μελών. Τι σχέση λοιπόν έχει το σύστημα αυτό και ε, το σύστημα ασφαλείας. Υπάρχει τέτοια σχέση, διασφαλίζεται για το μέλλον. Και τρίτον, σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε ήδη επικοινωνία G2, G3, G4. Δεν είχα το χρόνο να διαβάσω την μελέτη που μας ε, υποβάλατε, αλλά θα παρακαλούσα να μας απαντήσετε σύντομα στις ερωτήσεις αυτές. Η κυρία Μάισνερ, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Η κυρία Μπιλπάου είναι ε, ειδική στη διαλειτουργικότητα, τα περισσότερα λοιπόν θα τα αφήσω σε αυτήν. Αλλά στην ε, Γερμανία υπήρχαν προβλήματα, στη Βαβαρία είχαν προχωρήσει πολύ τα ε, πράγματα, αλλού όχι. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Λίθενμπεργκερ. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτηση του κυρίου Γκρός, διότι αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Το είχαμε συζητήσει αυτό στην Επιτροπή μας. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα τις ενδεχόμενης εφαρμογές διαφορετικών συστημάτων ε, για να, ε, ε, και να δυσκολεύσουμε έτσι την πρόσβαση στην αγορά. Έτσι όμως τελικά το σύστημα αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει πράγματι να έχουμε συνεχώς νέα συστήματα. Έτσι δίνουμε σε κάποιους σιδηρόδρομους τα μέσα να κάνουν διακρίσει. Πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό και να μην είμαστε αντιπαραγωγικοί. Και όσον αφορά την συγχρηματοδότηση για το τροχαίο υλικό, γιατί, προχωράει το θέμα, γιατί δεν προχωράει το θέμα αυτό, τι μορφή έχει το πρόγραμμα και να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Γκρός. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης ε, της ε, Συνδρομικής Πληροφορίας αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Στην ε, Αυστρία, στις Άλπεις, όπου ήδη έχει εφαρμοστεί το θέμα αυτό, πολλοί ιδιώτες, ε, πολλοί ιδιωτικοί φορείς δεν έχουν εφαρμόσει το σύστημα αυτό, δεν ε, περνάνε μέσα από το τούνελο που υπάρχει το ERMTS. Έτσι λοιπόν περνούν από κατοικημένες περιοχές με πολύ θόρυβο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εφαρμόζονται παράλληλα τα δύο συστήματα αυτά. Και αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Ε, τα, τα κράτη ε, επενδύουν τεράστια ποσά για κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά, διότι δεν είναι κατάλληλο το τροχαίο υλικό. Και τελικά δεν μπορούμε να φροντίσουμε οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτήν την υποδομή που δημιουργήσαμε για να είμαστε τεχνικά επικαιροποιημένοι, για να μειώσουμε το θόρυβο, για να εξυγχρονιστούμε. Δεν εφαρμόζεται λοιπόν το σύστημα αυτό λόγω των καθυστερήσεων στι επενδύσει. Γι' αυτό για μένα αποτελεί βασικό πρόβλημα και θα ήθελα να ξέρω τι λύση προτείνεται γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις εξηγήσει. Θα αναλύσουμε φυσικά την έκθεση με τη δέουσα προσοχή. Αλλά θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα εγκρίναμε την έκθεσή μας για τη διαλειτουργικότητα. Αφορά το τεχνικό πυλώνα του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου. Και μετά από εργόδεις προσπάθειες και επίπονες διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε ότι για τις, ε, η ΕΡΑ θα είναι η αρμόδια για τις άδειες του RTMS και μετά από διαβούλευση με τους εθνικούς φορείς. Φαίνεται όμως ότι το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη θέση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τις θετικές πτυχές που μας απαριθμίσατε και καλά κάνατε, εγώ συγκράτησα ένα πολύ σημαντικό θέμα ένα σημαντικό πρόβλημα, την ανομοιόμορφη ε, εξέλιξη. Δηλαδή κάθε μία από τις εθνικές ε, υπηρεσίες ε, θα, τραβήξει το δρόμο, θα τραβήξει δρόμο της. Και η έκθεση για τη διαλειτουργικότητα αυτό το πρόβλημα προσπαθούσε να διορθώσει. Αν λοιπόν το Συμβούλιο δεν συμπαραταχθεί με την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύετε ότι θα είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τις καλοπροαίρετες μεν ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, που όμως μάλλον αναποτελεσματικές θα είναι. Είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας των Σιδηροδρόμων είναι ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζουν 36 ε, χώρες στον κόσμο και το μιμούνται. Κάτι που σημαίνει ότι ως Ευρωπαίοι μπορούμε να αναπτύξουμε μοντέλα που θα γίνουν παγκόσμια σημεία αναφοράς. Μετά όμως από την παρατήρηση, την, παρα... την παρουσίαση που μας κάνατε, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο από όλα τα μοντέλα. Γιατί δεν υπάρχει ένα μόνο ενιαίο σύστημα ERTMS. Εγώ είμαι από τη χώρα των Βάσκων, αλλά στην Ισπανική κυβέρνηση, στην Ισπανική επικράτεια έχουμε ένα σύστημα ERTMS που μπορεί να είναι και ασύμβατο με τα αντίστοιχα άλλα συστήματα διαχείρισης τη κυκλοφορία, των σιδηροδρόμων. Επίσης μιλούμε για το υπέρογκο κόστο αυτή τη ανάπτυξη ε, των μοντέλων. Ποιο θα είναι λοιπόν το ευρωπαϊκό μοντέλο που θέλουμε να το εξαγάγουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Και επίσης ποιο θα είναι το κόστος ε, αν κάθε εθνική αρχή, κάθε εθνική υπηρεσία τραβήξει το δρόμο της και κάνει ε, το δικό της. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Αρχή με τις αρμοδιότητες ε, που έχει λάβει θα μπορέσει να διαχειριστεί, να κάνει το διαιτητή στην κατάσταση αυτή. Αν ε, οι χώρες δεν δεχτούν την ιδέα να γίνει ο συντονισμός ε, του σχεδίου αυτού σε κεντρικό επίπεδο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, γιατί εκεί έγκυται το πρόβλημα. Τα τεχνικά προβλήματα θα τα επιλύσουμε. Τα οικονομικά, αν υπάρξει πολιτική βούληση, επίσης θα τα ξεπεράσουμε. Υπάρχει όμως πολιτική βούληση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν θέλουν να εκχωρήσουν αυτή την αρμοδιότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Και σίγουρα το πρόβλημα εδώ είναι πολιτικό και όχι τεχνικό. Ερωτώ λοιπόν. Με μια τέτοια θέση του Συμβουλίου πιστεύετε ότι θα ευοδοθούν οι ωραίες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα συνεχίσω να υπερασπίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη... τις προσπάθειές του, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο ε, μοντέλο ευρωπαϊκό που θα μπορέσουμε να το προτάξουμε και ως ε, παράδειγμα προς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά δυστυχώς τα πολιτικά προβλήματα και μια κοντόφθαλμη αντίληψη που έχουν τα κράτη-μέλη για την πρόσπιση των εθνικών του συμφερόντων ίσως μας κάνει να χάσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να γίνουμε πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και σημείο αναφοράς. Ευχαριστώ κύριος Μπάνιον. Αναφερθήκατε στα θέματα ορισμένων περιοχών όπου το θέμα της χρήσης δεν έχει μόνο οικονομική ε, διάσταση. Ξέρετε γιατί η κίνηση, μιλάμε γιατί επίπεδο κυκλοφορίας ε, πρέπει να μιλάμε ε, όταν μιλάμε για αυτοχρηματοδότηση ή εκεί που χρειάζεται επιδότηση. Και ξέρετε πώς έχει η ε, κατανομή αυτών των μη ε, οικονομικά επικερδών ε, οδικών αρτηριών και μάλλον σιδηρομικών αρτηριών και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εξελιχθούν. Τσίκαου. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή το εξής. Ξέρουμε ότι η νομοθεσία που έχει εγκριθεί για το σιδηροδρομικό πακέτο, όχι δηλαδή στην τελευταία του έκδοση αλλά την προηγούμενη, σε αυτό το πακέτο υπήρχαν διευκολύνσεις σε σχέση με την πρόσβαση στην υποδομή αν τα τρένα ε, έχουν και χρησιμοποιούν το σύστημα ERTMS. Μπορείτε να μας πείτε τι επενδύσεις έχουν γίνει έτσι ώστε έμπρακτα να υπάρχει διευκόλυνση στη χρήση υποδομής των τρένων που διαθέτουν το ERTMS. Και ιδιαίτερα το σύστημα τροχοπέδησης ε, τη στιγμή που το τρένο ξεπερνά την ορισμένη ταχύτητα. Ξέρω, γνωρίζω ότι το ατύχημα της Ισπανίας θα είχε αποφευχθεί εάν η περιοχή αυτή ε, διέθετε το ETCS, δηλαδή το σύστημα τροχοπέδησης και θα ήθελα να μας πείτε πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε και τη χρήση αυτού του συστήματος ε, τροχοπέδησης. Πρόεδρος, κύριο Σε σχέση με το ε, τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και τον τεχνικό πυλώνα, θα ήθελα να πω κατά πόσο, να ρωτήσω κατά πόσο η Επιτροπή μπορεί να πείσει την Ιταλική Προεδρία να προωθήσει την ενιαία διαδικασία αδειοδότησης του ERTMS. Πολλοί έθιξαν το σύστημα αυτό G3, G4, αυτό το σενάριο. Και σε σχέση με τις δοκιμές και τις προδιαγραφές δοκιμών, που δεν είναι ε, έτοιμες. Η έκδοση 3.3 θα υποβληθεί στην Επιτροπή τον Ιούνιο. Άρα ε, στέλνουμε την τρίτη έκδοση στην Επιτροπή τον Ιούνιο, αλλά τώρα εργαζόμαστε επί μίας νέας έκδοσης 3,4 ε, πέρα από τις ε, δοκιμές. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε μία ε, έκδοση η οποία θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα. Γιατί ως προς τις ε, δοκιμές αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Και αυτά που είπε, αυτό που είπε η κυρία Μπιλμπάου για τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη δεν δέχονται με ανοιχτές αγκάλες αυτό το project. Δεν έχει σχέση με τεχνικά ζητήματα ή σιδηροδρομικά, αλλά καθαρά πολιτικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές. Ε, όσες φορές θέλουν και το κάνουν. Είτε θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ή δεν θα το, θα το διαθέσουμε, δεν θα το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, εντάξει, ε, ας επανέλθουμε στο αρχικό μας σχέδιο, αλλά αν διαθέτουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, τότε θα πρέπει να είναι πραγματικά ενιαίο. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν παρεκκλήσεις. Και θα ήθελα να υποβάλω και δύο άλλες ερωτήσεις τεχνικής υφής. Γιατί τα σημεία επαφής του ε, ERTMS και άλλων ε, συστημάτων όπως η, ε, η τροχοπέδηση γιατί δεν περιλαμβάνεται στο CCS ή στα άλλα η ETSI. Μου φαίνεται παράλογο, παράλογη η μη συμπερίληψη. και γιατί μπορεί κανείς να εισάγει το ERTMS από έναν κατασκευαστή τη στιγμή που πρόκειται για ε, ένα ενιαίο σύστημα. Γιατί ε, δεν ε, λειτουργεί το σύστημα ERTMS e όταν ε, εισαχθεί από έναν κατασκευαστή αλλά χρησιμοποιεί τροχαίο υλικό ενός άλλου κατασκευαστή. Γιατί δεν υπάρχει συμβατότητα. Πολύ σωστά ορίσατε τα προβλήματα, το πρόβλημα τεχνικής υφής και το οικονομικό σε σχέση με το τροχαίο υλικό στα κράτη-μέλη, αλλά ως προς την ε, τεχνική πτυχή ε, ορίσατε πολύ καλά τον πολυσχηδή της χαρακτήρα. Για μένα και τον Πατρίτσιο που εργαζόμαστε ε, σε καθημερινή βάση στον οργανισμό, ε, θέλουμε καταρχήν να παγιώσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, διότι αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα σχέδιο όπου κάθε δύο μήνες υπάρχουν νέες προδιαγραφές, τότε δεν καταλήγουμε πουθενά. Άρα η απάντηση βρίσκεται στο μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου, αυτού που υποστηρίξετε, που δυστυχώς δεν έτυχε υποστήριξης από το Συμβούλιο και αναμένουμε τις επικείμενες διαπραγματεύσεις των δύο συνομοθετών και θα πρέπει ο οργανισμός να είναι υπεύθυνος όχι μόνο για την πιστοποίηση του τροχαίου υλικού, αλλά και για την πιστοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Και η αρμοδιότητα του οργανισμού ε, βασίζονται στο γεγονό ότι θα είναι η ενία και μοναδική αρχή για την έγκριση του συστήματος ERTMS. Αυτό είναι αναπόδραστο στοιχείο, αν θέλουμε το σύστημα να είναι λειτουργικό. Προσπαθούμε να προβλέψουμε για τις άλλες αρμοδιότητες του οργανισμού. Θα θέλαμε ο οργανισμός να είναι πιο αυστηρός από το παρελθόν, δηλαδή να προετοιμάζει το έδαφος για την τελική ψηφοφορία της Επιτροπής τον Ιούνιο σε σχέση με τη βάση εργασίας της έκδοσης 3,3, Δηλαδή, το σύστημα θα βελτιωθεί, αλλά με αυτή τη βάση. Άλλοι μιλάνε για νέες εκδόσεις 3, 4, 3, 5. Βεβαίως θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την ε, ε, βελτίωση του συστήματος, αλλά υπό τον όρο ότι υπάρχει η εγγύηση της συμβατότητας, της προγενέστερης συμβατότητας και τα νέα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν με βάση την έκδοση Τρία-τρία που είναι και η έκδοση αναφοράς. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει η πειθαρχία του τομέα. Εδώ επήλθε μία σημαντική αλλαγή περιγράψατε ορισμένα προγρήματα με τον εξοπλισμό που θα πρέπει να τύχει προστασίας στο δίκτυο για να προστατεύσουμε την αγορά. Η βιομηχανία συνειδητοποίησε ότι θα πρέπει να ταχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να είναι ανοιχτή σε λύσεις. Και αυτό το είδαμε στην προετοιμασία μετάβασης στο σιδηροδρομικό σύστημα Δηλαδή η βιομηχανία ενδιαφέρεται για, το, για την πτυχή της διαλειτουργικότητας. Και με βάση το, την έκδοση 3.3 βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πειθαρχία και από τους φορείς και από τη βιομηχανία. Ε, εκεί που θα πρέπει να σταθούμε ε, αφορά τις εθνικές αρχές ασφαλείας γιατί υπάρχουν ε, αρχές που πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δεν έχουμε ακόμα το τέταρτο πακέτο, άρα μπορούμε με τη βοήθεια των συντονιστών και της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σίδηροδρόμων να τους ε, πείσουμε για την αξία ορισμού των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στις οποίες θα πρέπει να σταθούμε και να προβλέψουμε και βελτιώσεις για το μέλλον υπό τον όρο ότι θα είναι συμβατές με τη λύση που προβλέπουμε, το 3-3. Γι' αυτό είμαστε και αρκετά αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε, γιατί σε τελική ανάλυση όλοι αναγνωρίζουν ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει ε, στις διάφορες, στα διάφορα μέρη της Ευρώπης δεν θα έχουν νόημα αν το σύστημα λειτουργεί ανομοιόμορφα και έχουμε ένα ψηφιδωτό διαφορετικών συστημάτων. Τώρα, στα θέματα της επικοινωνίας. Φυσικά εξετάζουμε πολύ σοβαρά τα θέματα των παρεμβάσεων. Σε μερικά σημεία του δικτύου, εξαιτία ε, της ε, μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού, μερικοί υπάρχοι τηλεπικοινωνιών ε, δίνουν περισσότερη ενέργεια και υπάρχουν κάποιες παρεμβολέ. Δεν είναι τεχνικό όμω το πρόβλημα, ευτυχώ. Ευτυχώς δεν είναι ακόμη ένα άλλο τεχνικό θέμα, ένα άλλο τεχνικό εμπόδιο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Απλώς θέλουμε να βάλουμε μια επιθαρχία στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για να ευθυγραμμιστούν με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ενέργεια. Το όριο που θα πρέπει να τηρήσουν. Τελεία και παύλα τίποτα παραπάνω. Αυτό θα το δούμε με τους συναδέλφους για τη διαχείριση του φάσματος ε, και με, τους, ε, με τις ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό το έχουμε ήδη κάνει. Αναφερθήκατε στην ε, απαραίτητη εξέλιξη του συστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Σιδηροδρόμου προς τη νέα γενιά των τηλεπικοινωνιών, Τρίτη γενιά και τέταρτη γενιάς. Αλλά όχι τώρα παρακαλώ, για να μην καθυστερήσουμε το όλο θέμα των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών. Θέλουμε καταρχήν κάτι που να λειτουργεί παντού, εύρυθμα και μετά σταδιακά, προοδευτικά θα εξετάσουμε τις περαιτέρω βελτιώσεις. Και η απαραίτητη φυσιολογική μεταστροφή προ τρίτη και τέταρτη γενιά θα γίνει, αλλά πρώτα θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ε, με σωστές ε, τεχνικές προδιαγραφές με τις ισχύουσες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Μας επισημάνατε κάποιες δυσκολίες στη Γερμανία. Στις περισσότερες χώρες έχουμε πραγματικά μεγάλη δέσμευση. Το γερμανικό ζήτημα έχει επιληθεί πολύ δύσκολο και ήταν από τα βασικά επιτεύγματα πέρυσι του Κάρλ Ελβιν ότι βρήκε λύση που έπεισε όλους τους ενδιαφερόμενους στη Γερμανία, ακόμη και τους Βαβαρούς, για να συνεχίσουμε το ERTMS παράλληλα με τις προτεραιότητες που έχουμε για τους διαδρόμους ε, ERTMS και τους διαδρόμους ε, μεταφορών εμπορευμάτων. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα και καταπληκτικό του Ηνωμένου Βασιλείου Εκεί ήταν πολύ επιφυλακτική απέναντι στο RTMS αρχικά, αλλά χθε ανήγγυλαν ότι θα το εφαρμόσουν σε όλη τους την επικράτεια. Οπότε το μόνο να απομείνει σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ένα. Το συζητούμε και προσπαθούμε σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουμε τις σωστές προτεραιότητες, ώστε βραχυπρόθεσμα να καλύψουμε όλα τα κενά ακόμη και στο θέμα των συνόρων αυτό που επισήμανε δηλαδή η κυρία Λίχτεμπεργκ. Τώρα, τι εξουσία έχουμε απέναντι στα κράτη-μέλη και στους διαχειριστές υποδομών που σε τελική ανάλυση είναι αυτοί που θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμη το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, το, η μόνη εξουσία που έχουμε, η μόνη ισχύς που έχουμε είναι η ισχύς της πυθούς. Προσπαθούμε δηλαδή να αποδείξουμε την αξία του συστήματος και φυσικά Θέλουμε να εφαρμοστεί το νέο σύστημα για να αντικατασταθεί παροχημένη τεχνολογία ή να ισχύσει το ERTMS εκεί που επιτρέπει οικονομίες, γιατί πραγματικά γίνονται σοβαρές εξοικονομήσεις. Επίσης θα θέλουμε καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές, ώστε να επικεντρώσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Και κάτι που αναφέρετε κι εσείς, δεν έχουμε ήδη έτοιμες λύσεις ε, για τη χρήση του RTMS και της, ε, την πρόσβαση στην κατανομή των, ε, του κόστους. Υπάρχει ήδη στην αναδιατύπωση. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη των επιπτώσεων, οπότε ελπίζουμε φέτος να υποβληθεί η πρόταση, αλλά θα χρειαστεί χρόνος μέχρι ότου εφαρμοθεί. Θα πρέπει πάντως οι διαχειριστές υποδομών να καταλάβουν ότι το RTMS δεν θα είναι μόνο κόστος, αλλά θα εξασφαλίσει και έσοδα. Γιατί όσο περισσότερο RTMS έχουμε, τόσο περισσότερα εμπορεύματα θα κυκλοφορούν στις σιδηροδρομικές τους γραμμές. Σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, έχουμε ήδη περιλάβει στο έγγραφο ένα χάρτη της Ευρώπης με τα κενά που υπάρχουν Τώρα, για τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουμε ακόμη τις προβλέψεις, είναι πιο περίπλοκη κατάσταση, θα εξαρτηθεί από το είδος της κυκλοφορίας και το τι κυκλοφορία θα δημιουργηθεί περαιτέρω με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της θέσης μου εδώ, της ιδιότητάς μου ως αλλά το θέμα της επαφής, της διαπαφής του ARTMS με άλλες σιδηροδρομικές λειτουργίες γιατί είπατε ότι είναι έτοιμο το σύστημα και τα έγγραφα το τεχνικό προδιαγραφών είναι έτοιμα και η ε, Επιτροπή Αρμόδια έχει συμφωνήσει με τη συμπερίληψη, αλλά πού έχει κολλήσει το πράγμα. Γιατί μιλήσατε για το σύστημα της τροχοπέδης και της, ε, τη διασύνδεση με αυτό και είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Τι συμβαίνει ως προς αυτό το σημείο. Πρόκειται για ένα θέμα που το εξετάζουμε. Ο οργανισμός ε, το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τα τεχνικά, τις τεχνικές πτυχές του ERTMS γιατί όσο περισσότερες απαιτήσει έχουμε, τόσο πιο περίπλοκη γίνεται τεχνικά η κατάσταση και τόσο μεγαλύτερη καθυστέρηση έχουμε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τεχνικών χαρακτηριστικών. Θέλουμε όλα αυτά να είναι έτοιμα μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να μπορέσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να επιταχύνει τις εργασίες και να μπορέσουμε να δώσουμε και μια θετική απάντηση στο εύλογο δικό σας θέμα, γιατί μέχρι στιγμής ε, θεωρήθηκε ο οργανισμός ότι λειτουργούσε εν κενό, ενώ ουσιαστικά θέλει να, δημιουργήσει, να ε, προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστημα. Το βασικό ζητούμενο όμως εδώ είναι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μετά θα δούμε τη διασύνδεση με τα άλλα χαρακτηριστικά στο σειρμό, τις νέες τεχνολογίες ε, τηλεπικοινωνιών, τις τεχνολογίες νέας γενιάς και ούτω καθεξής. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η τυποποίηση έχει συμφωνηθεί. Είναι έτοιμα τα σχετικά έγγραφα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή του ERTMS έχει συμφωνήσει. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν διαφωνίες στο θέμα αυτό. Γιατί λοιπόν όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ναι, έχει συμφωνηθεί η τυποποίηση αλλά θέλω να υπάρχει πρώτα ευρωπαϊκή προδιαγραφή και μετά θέλω να εξετάσω τις ε, περαιτέρω πιθανές βελτιώσεις του συστήματος. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά τις εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή πάλι, ε, συγγνώμη, υπάρχουν τεχνικά πρότυπα, αν τα εφαρμόσουμε θα ε, καθυστερήσουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί. Η κυρία Λίχτερμπέργκερ. Μία παρατήρησή μου δεν απαντήθηκε. Έχουμε σημαντικά προβλήματα σε αυτή την διαδρομή βορρά-νότου. Οι δημόσιες εταιρείες έχουν κάνει τις προσαρμογές του τροχαίου υλικού, οι ιδιωτικές όμως όχι. Θέλουμε όμως ε, τα τρένα να ακολουθούν αυτή τη διαδρομή και όχι να ακολουθούν ε, εναλλακτικέ διαδρομές. Κάθε επένδυση λοιπόν ενός κράτους που θέλει να εφαρμόσει το σύστημα αυτού χάνει το νόημά της εάν τελικά το σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή κάποιες ιδιωτικές εταιρείες αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτά τα προβλήματα, διότι κάποια στιγμή χάνονται έτσι και τα κίνητρα. Έχουμε στην Βιέννη εν μέρη το σύστημα αυτό. Έχουμε στο σημείο που συνορεύουν τρεις χώρες, αλλά πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε απέναντι στους φορολογούμενους τις συνεχείς επενδύσεις στο σύστημα αυτό εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή ακριβώς ε, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θέλουν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό. Δεν έχω ακόμα το πακέτο ώστε να μπορέσω να προσφύγω κατά αυτών των εταιριών, αλλά ο κύριος Βίνκ μπορεί να πείσει τις αρμόδιες αρχές ε, να επιβάλλουν περισσότερη πειθαρχία στις ιδιωτικές εταιρείες και σίγουρα να μην παρέχουν δημόσια χρηματοδότηση σε όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες. Δεν μπορώ όμως να προσφύγω εναντίον του στο δικαστήριο, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ακόμα μηχανισμό επιβολής των κανόνων αυτών. Ακόμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αρκετά τεχνικό το ζήτημα, είναι όμως και πρόβλημα που εγείρει πάθη. Στους σιδηροδρόμους πάντα φαίνεται να κολλάνε τα πράγματα. Και ξέρω ότι οι ευρωβουλευτές νιώθουν μεγάλη δυσαρέσκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ όμως για την αναφορά σας. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Βίνγκ. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις προσπάθειές του όσον αφορά τους ε, σιδηροδρόμους. Έχουμε ε, προσκεκλημένου ε, κάποιου δημοσιογράφου από την εκλογική περιφέρεια τη κυρία Ετικάου. Παρ' όλα αυτά, θέλω, παρότι φτάνουμε στο τέλο τη ε, συνεδρίασή μα, θα ήθελα να του καλωσορίσω. Δεν έχουμε θέμα, κανένα θέμα στα διάφορα. Η ημερομηνία τη επόμενη συνάντησή μα που θα είναι η τελευταία τη επιτροπή μα κατά τη διάρκεια αυτής της θητεία, θα είναι 5η-10 Απριλίου στι 9 το πρωί. Τζαν 6Q2 θα είναι η αίθουσα. 6Q2 λοιπόν, 10 Απριλίου, 9 η ώρα το πρωί είναι η τελευταία μας ε, συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ ε, όλους.